από τους μεγαλύτερους ευρωπαίους εξαγωγές και τους μεγαλύτερους ευρωπαίους εξαγωγείς νερού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί για δύο μισή λεπτά από την ομάδα των Φιλελευθέρων και, μετα... και Δημοκρατών ο κύριος Καζάκ.